Welcome everybody to the Budget Committee meeting. Uh, first point. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Πρώτο σημείο με έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις του Προεδρού, αποφάσεις των συντονιστών από τις 30 Σεπτεμβρίου του 2019 μπορούν να βρεθούν μεταξύ των φακέλων σας, των εγγράφων σας. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνονται και αυτές. Και τρίτον, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων και πάλι ε, συνεδρίαση για τις 14 Οκτωβρίου του 2019. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνονται και αυτά. Περνάμε τώρα την ψηφοφορία. Καταρχάς, η Συμφωνία Βιώσιμης Αλίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπια και της εφαρμογής ε, του σχετικού πρωτοκόλου. Να κάνουμε μια δοκιμή καταρχάς ε, για τα μηχανήματα, για να δούμε ότι λειτουργούν όλα όπως πρέπει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Όχι. Ψήφισαν όλοι. Ωραία, πέρασε τη ψηφοφορία. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, αλλά από ό,τι φαίνεται λειτουργεί. Το πρώτο σημείο λοιπόν είναι αυτή η συμφωνία για την αλία που μόλις σας ανέφερα. Ψηφοφορία μονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις ενημορήθηκα ότι το Συμβούλιο απέρριψε αυτή τη πρόταση για του Ταμείου, του Κινητοποίηση για την Παγκοσμιοποίηση, για τους ανθρώπους που έχασαν τις θέσεις εργασίας τους, θύματα της παγκοσμιοποίησης. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αντίστοιχες, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και είναι απαράδεκτο ε, να έχουμε τέτοια στάση από το Συμβούλιο. Πρόκειται για κάτι που καταδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών είναι ανύπαρκτη και αυτό φυσικά θα πρέπει να μας ανησυχεί και υπάρχει και το εξή. Το ταμείο αυτό, το οποίο είναι για εργαζομένους, για ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τις θέσεις εργασίας τους, ε, οι περισσότεροι από, είναι, αυτούς είναι άνω των 55 ε, ή πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης και θα βρεθούν και αυτοί άνεργοι και το Συμβούλιο χωρίς καμία αιτιολόγηση δεν εγκρίνει αυτή την ε, πρόταση όπως είχε κάνει στο παρελθόν για αντίστοιχες περιπτώσεις. Οι κανόνες για το επόμενο Ταμείο Προσαρμογής της ε, Παγκοσμιοποίησης, αν θέλει να τους αλλάξει το Συμβούλιο, αφορούν το μέλλον δεν μπορεί να αλλάξει τους κανόνες ε, για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ε, για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να τα αλλάξει, και, αλλά αρχίζει να τα εφαρμόζει ήδη από τώρα. Βάσει των κανόνων που έχουμε τώρα, το Συμβούλιο θα πρέπει να διαβάσει και να εξετάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αντίστοιχη με άλλες προτάσεις. Γι' αυτό λοιπόν να πω ότι η θέση του Συμβουλίου είναι επονίδιστη και δεν σέβεται τους κανόνες, το δίκαιο και φυσικά τους Βέλγους πολίτες που έχασαν τις ε, δουλειές τους σε μια περιοχή όπου ε, ε, το ποσοστό της ανεργίας είναι διπλάσιο από άλλες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, θα ψηφίσουμε τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ή μάλλον, καταρχάς, τροπολογία 2. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπολ 10, καταπίπτει, τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. 6. Την 6 ψηφίζουμε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπολ 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην αιτιολογική σκέψη ε, ε τροπολογία 1, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του εγγράφου με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με 30 ψήφους υπέρ και 3 κατά. Ο κύριος ε, Σαστέλ θέλει να σχολιάσει κάτι για τις ψηφοφορίες. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, προφανώς και θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πολύ σημαντική αυτή ψηφοφορία και επίσης ε, να Χαιρετήσω την αποφασιστικότητα του εισηγητή μας, ε, διότι ευθύς εξ αρχής ε, εργάστηκε με συνέπεια ε, για τα όσα έγιναν στο θέμα αυτό και για συγκεκριμένη νομολογία η οποία ήταν αυτή η οποία ήταν δεσπόζουσα στις περιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Δεν θα επισέλθω στην ουσία, είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζω καλά. Είναι ένα θέμα το οποίο άφησε στο δρόμο αρκετούς εργαζομένους και μέχρι τώρα έχει αποδείξει όλη την ε, ε, προστιθέμενη αξία του και πώς μπορούμε να αντισταθμίσουμε τις συνέπειες της ε, παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης. Μέχρι τώρα λοιπόν ήταν προστιθέμενη αξία να αποδείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παρέμβουν να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Ο εισηγητή το κατάλαβε, έχει εμπειρία στον αυτό και τον ευχαριστώ. Και συμφωνώ απόλυτα με τη δήλωση της χώρας μου, του Βελγίου, ε, στις διάφορες συνεδριάσεις του Συμβουλίου, είτε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, είτε ε, στον τρόπο ε, με τον οποίο η Αντίτσι και σήμερα το πρωί η Κορεπέρ, το Βέλγιο, είπε ότι λυπάται για αυτή την απόφαση. Μόνο μία χώρα καταψήφισε αυτή την πρόταση. Πολλές χώρες απήχαν δεν υπήρχε λοιπόν ε, ειδική πλειοψηφία για να εγκριθεί η πρόταση στην Κορεπέρ και θα πάμε σε ένα τριμερή διάλογο όπου ε, πραγματικά το περιθώριο λιγμών είναι πάρα πολύ περιορισμένο και λυπάμαι για αυτό το προηγούμενο. Και όπως και ο εισηγητής, λυπάμαι κυρίως όπου το Συμβούλιο φαίνεται ήδη να έχει αρχίσει να σκέφτεται την εξέλιξη των διαφόρων εξετε, ε, περιπτώσεων κινητοποίηση του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση, ενώ εδώ θα έπρεπε να βασιζόμαστε στους κείμενους κανόνε. Αυτά θα ήθελα να πω ω τελική δήλωση. Ωραία, περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Μακροοικονομική συνδρομή στο χασεμητικό βασίλειο της Ιορδανίας. Έχουμε μια επιστολή για το θέμα αυτό, η οποία έχει διανεμηθεί και έχουμε μια τροπολογία των σοσιαλιστών και δημοκρατών η οποία έχει συμπεριληφθεί και έχει εγκριθεί από τους ε, συντονιστές στην ε, συνεδρίαση που κάναμε προηγουμένως. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο τμήμα 3 του 2019 και να δώσω το λόγο στον κύριο Χάουερθ, τον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρώτη από αυτές τις μεταφορές ε, σήμερα, 18, έχει να κάνει με την προσαρμογή, το Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο μόλις εγκρίνεται. Η μεταφορά έχει να κάνει με 1.632.028 ε, άμα από τη γραμμή 40.0243 και θα ήθελα να κοιτάξουμε τον κανονισμό ε, λεπτομερώς ό,τι αφορά το νέο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο θεωρώ ότι θα περάσει και στο νέο προπολογισμό. Δεν μιλάμε μόνο για το πρώτο τμήμα. Και γιατί με απασχολεί αυτή η μεταφορά. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι το θέμα αυτό θα περάσει στον τρομερή διάλογο, μεταφέρουμε το ποσό αυτό και θεωρώ ότι θέλουμε να πετύχει η μεταφορά αυτή. Θέλουμε λοιπόν να εγκρίνουμε το 10-18 ξεχωριστά. Για να υπάρχει σαφήνεια. Μάλιστα. Λέει ο πρόεδρο, θέλει κανεί να σχολιάσει από αυτού. Όχι. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Ζουρέλ, μήπω θέλει να πάρει το λόγο να σχολιάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να υποστηρίξω και εγώ α, αυτά που μα είπε ο κ. Φερνάνδε, ο κ. Αστέλ και ο κ. Χάουαρτ και να επιβεβαιώσω ότι θα μπει αυτό στην ημερήσια τέταξη του τριμερού διαλόγου για αύριο και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει το θέμα αυτό. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρο. Να περάσουμε στην ψηφοφορία. Όπω είπε και ο κύριο Χάουαρτ, να ακολουθήσουμε τη σύστασή του. Προτείνω να ψηφίσουμε ξεχωριστά το ΤΕΚ Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Το υπόλοιπα τεκ. Κύριε Χάουαρτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Να προτείνω τις άλλες μεταφορές να τις ψηφίσουμε από κοινού. Δεκ 20 μεταφορές 470.000 ε, ευρώ. από τις ε, ασφάλειες αγορών. Α, συγγνώμη. Προκειμένου να γίνουν δύο μελέτες για την εφαρμογή οδηγιών σε ό,τι αφορά τον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών και των ασφαλίσεων. Δεν 21 μεταφορές 100.000 ευρώ. 100 εκατομμυρίων για το Αφγανιστάν, Σαχέλ και το Σουδάν. ΔΕΚ 22. Διοικητικές μεταφορές σε διάφορους τομείς του ορίζοντα 2020 και σχετικών προϋπολογισμών. 3,3 εκατομμύρια σε δεσμεύσεις και πληρωμές. 10-23 μεταφορές ε, από τον Μηχανισμό Προστασίας Πολιτών στο σύστημα ασύλου και μετανάστευσης 45 εκατομμυρίων. 10-24 διοικητικές μεταφορές και πάλι. Από τον προπολογισμό για τα κτίρια στην πολιτική ανταγωνισμού 769.998 ευρώ. 10,25. Από το παθηματικό λοιπόν μεταφορές εδώ. 63,3 εκατομμύρια. Δεσμεύσεις. Και 54 εκατομμύρια 950.000 ε, δεσμεύσεις πληρωμών από τα παθηματικά στην πολιτική αλληλείας σε ό,τι αφορά συμφωνίε με την ε, Σενεγάλη και τη Μαυρετανία. Να προτείνω να τα ψηφίσουμε όλα αυτά μπλοκ. Ευχαριστώ κύριε Χάουαρτ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο να σχολιάσει. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι να προσθέσει. Όχι. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Α, συγγνώμη, θέλετε να πάρετε το λόγο, νόμιζα. Να ψηφίσουμε λοιπόν ένα μπλοκ. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Οι μεταφορέ λοιπόν για το 2019, τα υπόλοιπα τμήματα. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Φερνάνδη που είναι ο εισηγητή, θα ήθελα να εξηγήσω το εξή. Έχουμε δύο μεταφορές που σχετίζονται με το Brexit στην ημερήσια διάταξη, τις οποίες τις λάβαμε τη Δευτέρα μόλις. C15 που αντικαθιστά το C13 και το C16 λόγω της αναβολής ε, του Brexit ε, στον Ιανουάριο του 2020 και το Κοινοβούλιο λοιπόν θα χρειαστεί να κάνει κάποιε μεταφορέ δεδομένων των σημαντικών ζητημάτων λοιπόν, που μας ε, αντιμετωπίζουμε, αποφάσισα να μπουν κατά εξαίρεση αυτά τα θέματα στην ατζέντα, τα οποία δυστυχώ κατέφτασαν πάρα πολύ καθυστερημένα για την ιστορική μα διαδικασία. Κύριε Φερνάνδε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Λοιπόν, ε, για αυτή την παρουσίαση όλων αυτών των πιστώσεων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το C10 2019 αφορά τις ανάγκες τεχνολογικών υποδομών και έργα. Μεταβιβάζονται από τις δαπάνες για την κοινοβουλευτική συνδρομή. Έχουμε επίσης ε, τη γραμμή 24 ε, υποδομές 55.000 ε, ευρώ μέχρι προς την 2.105 ε, με όλες τις σχετικές πληροφορίες και μετά αυξάνονται οι δαπάνες που σχετίζονται με την επιπλέον συνδρομή 1.975.000 ευρώ. Μετά έχουμε την C11 αφορά προεκοδότηση της ε, διερμηνίας όπως προβλέπεται στον κανονισμό του Κοινοβουλίου σχετίζεται με τις δαπάνες ε, της διερμηνίας. Οπότε αυξάνονται οι δαπάνες για την διερμηνία κατά 1.800.000 ευρώ και μείωση της 42.20. Η αύξηση δηλαδή που έχουμε από τη μία πλευρά αντισταθμίζεται με τη μείωση στην άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία επίδραση στον ε, προπολογισμό διότι σωσταθμίζονται ε, δημοσιονομικά. Μετά το Κοινοβούλιο ζητά μια άλλη μεταβίβαση, την C12 του 2019, για να παράσχει περισσότερα κονδύλια για τις δαπάνες ε, που υπερβαίνουν τις αρχικές εκτιμήσεις. Μιλάμε για τις πολιτικές ομάδες τώρα που το συζητούν. Ειδικότερα αύξηση της 3042 κατά 300.000 ευρώ και μείωση της 2105 υπολογιστική και τα λοιπά αξίας 300.000 ευρώ. Για την C15 μόλις μίλησε ο πρόεδρος και για το ζήτημα του Brexit ε, αντικαθιστά την C13 αυτή η μεταβίβαση C15 αφορά τις δαπάνες που οφείλονται στην αναβολή του Brexit. Για τη γραμμή που αφορά μισθούς ε, και ε, αμοιβέ ε, υπάρχει προβλεπόμενη αύξηση. Και μετά για τις τακτικές δαπάνες 4.100.000 ευρώ και μετά αυξήθηκαν και οι άλλες δαπάνες αλλά οι δαπάνες αυτές αντισταθμίζονται από τη μείωση της γραμμής 1020 και μετά έχουμε μείωση επίσης και στην 1030 1.800.000 ευρώ και μειώνονται και οι δαπάνες κοινοβουλευτικών βοηθών 6.180.000 μείωση ε, τώρα το κοινοβούλιο για την ε, ε, ε, C16 προβλέπει και την καθυστέρηση του Brexit και εκεί προβλέπονται άλλες δαπάνες στην 32-42 προβλέπεται αξία ενό εκατομμυρίου 230.000 ευρώ και στην 32-44 για τους επισκέπτες και εκεί προβλέπεται αύξηση και στην 3248 δαπάνες ε, ε, οπτικοακουστικών πληροφοριών πάνω από ένα εκατομμύριο παραπάνω και 3250 δαπάνες για το Liaison Office 320.000 ευρώ. Πρόκειται για δαπάνες οι οποίες αντισταθμίζονται στην 3211 για παράδειγμα προβλέπεται αύξηση 650.000 ευρώ στην 1404 προβλέπεται μείωση των 176.000 ευρώ, μάθηση και ε, ανάπτυξη 150.000 ευρώ λιγότερα, στην 2026 ασφάλεια και φύλαξη κτηρίων, μείωση ε, κατά 1.330.000 ευρώ, 203 επικοινωνία και μείωση 330.000 ευρώ, 2020 ε, κόστος ε, για ε, νομικές ζημίες, επίσης μείωση και μετά για τους εμπειρογνώμονες έχουμε μία μείωση. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα προηγουμένως, όλες οι μεταβιβάσεις ίσως σταθμίζονται. Όσον αφορά το ελεκτικό συνέδριο, υπάρχει μεταβίβαση, αναφέρομαι στην C17 και C19 Έχουμε μεταβίβαση για το ελεγκτικό συνέδριο για ενίσχυση της 2102 εξωτερικές υπηρεσίες. για, την διατηρησή του, για τη συντήρηση του λογισμικού 340.000 ευρώ. Έξι μόνιμες θέσεις βοηθών θα γίνουν ε, διοικητικές θέσεις μόνιμες και αυτά τα 340.000 ευρώ αντισταθμίζονται με άλλες εξοικονομήσεις σε άλλες γραμμές του προπολογισμού. Επιτροπή των Περιφερειών 23-2019 ε, Έξι τομεί του προπολογισμού θα ενισχυθούν κτίρια και νέες τεχνολογίε, ειδικότερα συνολική μεταβίβαση 1.500.000 περίπου ευρώ. 1.519.000 ευρώ για την ακρίβεια για τη χρηματοδότηση συνολικά διαφόρων ανακαινήσεων, έργων πληροφορικής. Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται με εξοικονόμηση σε άλλα τμήματα του προπολογισμού ε, ΕΟ και έχουμε την μεταβίβαση 1-2019 ύψους 2.454.294 ευρώ. 1.400.000 ευρώ από αυτό το ποσό στις ε, καθυστερημένες πληρωμές ε, όσον αφορά τα κτίρια ε, για την περίοδο 2007-2008 και για την καταβολή για τις τεχνολογίες πληροφορικής. Μετά ζητείτε μεταβίβαση για μικρά έργα, μικρά, ε, μικρά εγχειρήματα. Οι μεταβάσεις αυτές έχουν ήδη γίνει δεκτές χάρη σε ε, εξοικονομήσεις που έχουν γίνει σε άλλα τμήματα του προπολογισμού. Όλες αυτές ε, οι μεταβιβάσεις έχουν διορθωθεί, εξεταστεί. Δεν μπορώ παρά να δώσω ευνοϊκή ψήφο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρτιζαβάλ, το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μας ε, δεν ε, θα έχει ένσταση για καμία από αυτές τις μεταφορές, αλλά μιας ε, που είμαι εγώ αρμόδια για αυτό τον θεαματικό κόσμο των μεταφορών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα από εδώ και πέρα, θα ήθελα να κάνω το εξή αίτημα. Όταν κάποιο διαβάζει τι πληροφορίε, ορισμένε φορέ δεν ξέρει τι διαβάζει. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Μια φράση λέει ο επιπλέον προπολογισμό θα καλύψει το συνολικό κόστος για την αγορά της ε, ε ενιαίας ε, άδειας Magic Shop. Δεν μπορεί κάποιο να είναι πυρογνώμων στα πάντα. Όταν μα δίνετε λοιπόν πληροφορίε για τι μεταφορέ, ε, να εξηγείτε λίγο και για του κοινού θνητού ε, για περί τίνο πρόκειται. Διότι σε κάποιε περιπτώσει ε, μπορούμε να τα εξηγήσουμε πολύ πιο εύκολα και μα διευκολύνει πολύ τη δουλειά μου και εμένα και την ομάδα μου που πρέπει να καταλάβουμε και γιατί συζητούμε. Και επίση και κάτι ακόμα. Σε πολλέ περιπτώσει και ε, εδώ δεν ξέρουμε, εδώ δεν υπάρχει, αλλά σε κάποιε άλλε περιπτώσει όχι. Ε, γιατί πρέπει να αιτιολογήσουμε τη συγκεκριμένη μεταφορά. Για παράδειγμα, στο Brexit ε, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχουν επιπλέον δαπάνε γιατί ευτυχώ οι Βρετανοί Ευρωβουλευτέ θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά σε ένα άλλο σημείο έχουμε αύξηση 50.000 ευρώ για αγορά εξοπλισμού πληροφορική και εκτυπωτέ για τα γραφεία των ευρωβουλευτών. Έχουμε τον ίδιο αριθμό ευρωβουλευτών, αυτό προβλεπό ε, το 2019 ούτως ή άλλως και ξέραμε ότι θα είχαμε διεύρυνση των γραφείων. Δεν ξέρω λοιπόν γιατί δεν είχε προβλεφθεί αυτό το επιπλέον κονδύλιο. Μπορεί γιατί δεν έφτασαν τελικά τα χρήματα και να θεωρήθηκε ότι η αγορά θα μπορούσε να γίνει αφού υπήρχαν, διαπιστωθεί ότι υπάρχουν επιπλέον κονδύλια. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ε, αν είχαν προβλεφτεί στον προπολογισμό κάποια πράγματα ή όχι. Επίση, ερώτηση όσον αφορά τους ε, κοινοβουλευτικούς βοηθού. Ερώτηση γιατί δεν ξέρω πώ λειτουργεί το θέμα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν ξοδεύουμε το 100%. Όλοι έχουμε διαθέσιμο κονδύλο και είναι δύσκολο να εκτελεστεί το 100%. Αλλά η ερώτησή μου είναι, είναι υποχρεωτικό να προβλεφθεί στον προπολογισμό στο 100%? Είναι απέτηση του προπολογισμού. Ορισμένε φορέ υπάρχουν τέτοιε απαιτήσει, υπάρχουν όλα αυτά τα χρήματα και πρέπει να ε, καταλογιστούν όλα. Και αν ε, ε, περισσέψουν μπορούμε να τα δώσουμε σε, σε άλλε ε, ε πτυχέ ή να τα μεταβάσουμε στην επόμενη χρονιά. Θέλω απλώ να ξέρω αν πρέπει να συμπεριληφθεί στον προπολογισμό στο 100%. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Κανεί άλλο από του κοιόδη εισηγητέ θα θέλει να πάρει το λόγο. Αν όχι. Ακούσαμε δύο επιχειρήματα ουσιαστικά από την κυρία μπαλ. Το πρώτο για τη σαφήνεια, το οποίο το υποστηρίζω απόλυτα. Ότι θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια. Και θα ήθελα να αναφερθώ να δώσω το λόγο μάλλον στον κύριο Πετρούτση για να μας ε, διαφωτίσει. Πού είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω, να σας δώσω πιο πολλές πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά τα θέματα των αδειών, το SAP αποτελεί ένα λογισμικό το οποίο χρειάζεται να αγοράσουμε για να διαχειριστούμε τους πόρους του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά το νέο οικονομικό, χρηματοοικονομικό σύστημα του Κοινοβουλίου συγκεκριμένα, προκειμένου λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να αγοράσουμε και τις σχετικές άδειε. Η άδεια συνεπάγεται δικαίωμα χρήσης του συστήματος. Χρειάζεται λοιπόν να αγοράσουμε κάποιες άδειες για να επιτρέψουμε σε όλους τους ενδυνάμει χρήστες του συστήματος να το χρησιμοποιήσουν όπως προβλέπετε. Αυτό λοιπόν περιλαμβάνει στο Κοινοβούλιο, στις διάφορες γενικές διευθύνσεις, προκειμένου να γίνει διαχείριση του προϋπολογισμού, ε, προβλέπεται εξειδικευμένο προσωπικό. Εξειδικευμένο για να διαχειρίζεται τα οικονομικά της Γενικής Διεύθυνσης και θα πρέπει να έχουν άδεια για να χρησιμοποιούν το λογισμικό αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να αγοράσουμε την άδεια αυτή. Πρόκειται για ένα μηχανισμό ο οποίος είναι ο κλασικός, θα έλεγα, στην, στο IT. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δεδομένου όμως της έκτασης της ε, εξήγησής σας, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν πιο σαφείς εξηγήσει και γραπτά, προκειμένου να καταλαβαίνει και ο κόσμος που δεν ε, είναι γνώστης. Για να καταλάβει δηλαδή ο καθένας τι αφορά αυτό το θέμα. Για το δεύτερο ζήτημα που έθεσε η κυρία Καρδία Ζαμπάλ, να δώσω το λόγο στον κύριο Μπάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Από τη Γενική Διεύθυνση Finance είμαστε και υπάρχει δικαίωμα το οποίο προβλέπεται του κανονισμό για κάθε βουλευτή που έχει βοηθούς. 24.000 είναι αναμήνα ο φάκελος αυτός. Για το τέλος λοιπόν του 2017, αρχές 2018, λαμβάνουμε υπόψη το συντελεστή εφαρμογής, υλοποίηση ε, που είναι κοντά στο 100% κάθε φορά. 2,8 εκατομμύρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αρκετά καλά. Προβλέπουμε λοιπόν στον προπολογισμό αυτό το ποσό. Τι έγινε τώρα στο έτος των εκλογών. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, δεν μπορούμε να προβλέπουμε τι θα γίνει. Για παράδειγμα, αυτή τη φορά είχαμε χαμηλό ποσοστό επανεκλογής των βουλευτών. Κυρίως είναι συνήθως γύρω στο 50%, τώρα ήταν στο 38%. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι βουλευτές πρέπει να βρουν ε, βοηθούς, να ξεκινήσουν ενδεχομένω με κάποιους ντόπιου. Και εδώ χρειάζεται λοιπόν πιο πολύ χρόνο για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Αυτό λοιπόν το ποσό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε άλλες ε, ανάγκες. Άρα υπάρχει μια βεβαιότητα ε, λόγω των ευρωεκλογών και λόγω του χαμηλού ποσοστού επανεκλογής των ίδιων βουλευτών. Ελπίζω έτσι να σας εξήγησα τι εννοούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπονφρίσκο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ιταλικά Πρόεδρε για να ζητήσω μία ε, εξήγηση από τον κύριο Πετρούτσι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς γίνεται αντί για κλασικές άδειες που δεσμεύουν, που σχετίζονται με τις αγορές λογισμικού και δεσμεύουν ε, το Κοινοβούλιο με διάφορες μονοπωλιακές, ε, πολυεθνικές στον κόσμο. Γιατί το Κοινοβούλιο δεν προσπαθεί λοιπόν να χρησιμοποιήσει Ε, να επαναχρησιμοποιήσει μάλλον ε, ε, άδειε που έχουν ήδη λάβει άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Κύριε Πετρούτσι. Thank you for this question. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Θα ήθελα να σας πω ότι η επιλογή της λύσης της ΣΑΠ από το Κοινοβούλιο έγινε μετά από διαβουλεύσεις ε, που έγιναν ε, ε, στην αγορά κυρίως από την EG από τον ιδιοκτήτη του έργου. Η EGI Tech φυσικά παρέχει την τεχνολογική υποστήριξη για τη λύση, αλλά τη διαβούλευση την κάναμε εμείς από κοινού με σύμβουλο, με εξωτερικό δηλαδή εξωτερική εταιρεία συμβουλευτικής υποστήριξης που εξέτασε τι ανάγκε, τι ιδιαιτερότητε του Κοινοβουλίου και βάσει αυτών πρότεινε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λύση. Φυσικά, εμεί μαζί με την Fins εξελογήσαμε ε, τις διάφορε διαθέσιμε λύσει ε, που υπάρχουν ήδη στα λαθισμικά όργανα αλλά δεν ήταν κατάλληλες για τις δικές μας ανάγκες. Και για τους εκτυπωτές. κοιτάξτε, κοιτάξτε μιλάτε για τους εκτυπωτές για τα μέλη. Ναι, πράγματι. Πρόσφατα αποφάσισε το Προεδρείο να παράσχει επιπλέον γραφεία στα μέλη. Στις κλασικές λοιπόν προμήθειες ε, για τα ε, μέλη παρέχουμε έναν ε, πολυλειτουργικό εκτύπωτη για κάθε μέλος και μετά υπάρχει και η δυνατότητα να αιτηθεί κάθε μέλος έναν επιπλέον εκτυπωτή για το άλλο γραφείο. Δεν είναι κάτι δηλαδή που γίνεται συστηματικά, αλλά μετά από έτοιμα. Αλλά πρέπει να αγοράσουμε κάποιον αριθμό εκτυπωτών για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των ε, μελών. Όχι μόνο εκτυπωτές, ε, αλλά επιπλέον γενικότερα υπολογισμό πληροφορική υπολογιστέ, ε, υβριδικά που είναι νέα κινητή λύση που παρέχουμε στα μέλη για να προωθήσουμε το ψηφιακό χώρο εργασία ε, που προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρο. Αυτή είναι μια τη μεγαλύτερη μεγαλύτερες που έχουμε κάνει ποτέ για μεταβίβαση, πιστεύω. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Σα ευχαριστώ όλου για τη συμμετοχή σα. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, οι μεταβιβάσεις C10, C11, C12 και C15 ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί. Και το ίδιο ισχύει, ε, κύριε Κούντς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ψηφίσω διαφορετικά. Ήθελα να ζητήσω τα... Ε, να ψηφίσουμε τα διάφορα σημεία αυτά ξεχωριστά. Ευχαριστώ. we will vote separately. So, C10. C10 λοιπον Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. C11. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία εγκρινεται Συ C12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. έκρινεται. C15. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Για το ελεγκτικό συνέδριο τώρα. Okay, we vote first on C. Να ψηφώσουμε πρώτα το C16. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Έγκρινεται. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, το ελεγκτικό συνέδριο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την ΕΟΚΕ μπορούμε να τις εγκρίνουμε αν δεν υπάρχουν στάσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι εγκρίνονται. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάτι για τα κτίρια στην ημερήσια διάταξη, επομένως ολοκληρώνεται εδώ η ψηφοφορία. Και περνάμε το σημείο 10, ανταλλαγή απόψεων για την, ε, το κτίριο Ζαμονέ στην πολύ ωραία περιοχή του Μπαζός. Κύριε Κέλλερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για προκοινοποίηση για ένα σχέδιο κτηρίου στο Μπαζός, στη Γιγιόμ, ε, σε ένα ιστορικό χώρο του Ζαμονέ να υπενθυμίσω εδώ ότι αγοράσαμε, ή τουλάχιστον οι προκάτοχοί μας αγόρασαν μία έκταση το 2018, 1.200 τετραγωνικά μέτρα για 250.000 ευρώ και πρόκειται για μία επιπλέον έκταση η οποία προτείνεται να ε, αγοραστεί. Υπάρχει και μια μικρή κατοικία εκεί και βρίσκεται ε, ακριβώς παρακείμενη στην έκταση ε, της οποίας είμαστε ήδη ιδιοκτήτες. Υπάρχει και ένα κέντρο διασκέψεων και το Μουσείο Ζαμονέ, διότι είναι το παλιο, η παλιά κατοικία του Ζαμονέ. Αλλά είναι όλα μικρά κτίρια. Δεν είναι κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, πρόκειται για μικρά, ε, μικρές μεζον, ε, μικρά σπιτάκια. Ε, η αγορά ε, προτείνεται λόγω ανάγκης για επιπλέον ε, ε, γραφεία, εκμετάλλευση του χώρου, ε, κατασκευή κατοικιών και βελτίωση της ασφάλειας. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω κάποιες ερωτήσεις ε, στις υπηρεσίες. Γίνεται αγορά έκτασης ε, από τον ίδιο ιδιοκτήτη από πέρσι, και πέρσι και γιατί δεν αγοράσαμε τα πάντα πέρσι, πρώτον. Δεύτερον, στην αιτιολόγηση αυτής της επιπλέον αγοράς υπάρχουν και θέματα ασφαλείας και ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Την ίδια ερώτηση έχω και εδώ. Δεν ε, τα ξέραμε αυτά πέρσι όταν έγινε αγορά του πρώτου τμήματος αυτής της έκτασης. Αυτά λοιπόν ε, αγαπητοί συνάδελφοι είναι τα ερωτήματά μου για το θέμα αυτά το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό από συμβολικής ε, σκοπιάς για τη ε, μνήμη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει κάποιος από τους Κιώδης να πάρει το λόγο, ο κύριος Κόζακοφς. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία, ε, μιας και έχουμε εδώ τις υπηρεσίες για να συζητήσουμε τα θέμα. Εγώ έψαξα στο Google που βρίσκεται αυτό το ιστορικό κτίριο και όταν διαβάζουμε ότι θα αυξηθεί ασφάλεια και θα αποφύγουμε αρνητικό αντίκτυπο από δραστηριότητε τρίτων, θα ήθελα να ξέρω το εξή. Το κτίριο βρίσκεται, είναι στη μέση του πουθενά. Τι θέματα ασφαλείας υπάρχουν ώστε να πρέπει να αγοράσουμε επιπλέον ε, γη. Επίσης, ε, Πήγα και στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ζαμονέ και στην ιστοσελίδα αναφέρεται η έκταση αυτή και θέλω να ξέρω κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εισοδήματα από αυτέ τι δραστηριότητε που προβλέπονται εδώ στην ιστοσελίδα και κατά πόσο η κατοικία, εφόσον είναι η ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί δεν έχουμε κάποια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ε, κέντρο Ζαμονέ. Ο κόσμο που τον νοικιάζει ξέρει ότι σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αρκούν αυτές οι ερωτήσεις για να καταλάβω γιατί χρειαζόμαστε να αγοράσουμε επιπλέον γη εκεί. Ο κύριος Αντρέσεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω δύο ερωτήσεις. Αν ο ιδιοκτήτης ήδη είχε κάνει προσφορά, ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας το πείτε δημοσίως, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον ε, να ξέρουμε αυτές τις πληροφορίες. Και έχω και μία ερώτηση για την κατάσταση της κατοικία ε, που βρίσκεται σε αυτή την έκταση γης. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν και ανακαινήσεις ή κάτι, κάποια άλλα έργα. Διότι αυτό έχει σημασία ως προς το κόστος. Είναι σημαντικές λοιπόν αυτές οι πληροφορίες. Άλλες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Ινλο και DGCOM. Να δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Μπαρ και στην κυρία Ιτσελ για να απαντήσω. Όποια θέλει μιλάει πρώτη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι η κυρία Μπάρα από τη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Λογιστικής σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρία Κέλλερ. Να σας πω ότι όντως ε, αγοράσαμε από τον ίδιο ιδιοκτητή φέτος το άλλο τμήμα της έκτασης. Προηγουμένως δεν μας είχε δώσει ο προσπόληση το άλλο τμήμα της έκτασης. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν μπορέσαμε να αγοράσουμε όλο το οικόπεδο την προηγούμενη χρονιά. Άλλαξε γνώμη στο μεταξύ και πλέον μας ε, προσέγγισε, μας είπε ότι θέλει να πουλήσει το σύνολο της έκτασης και να φύγει από εκεί και προφανώς θα θέλαμε να έχουμε αγοράσει όλη την έκταση εξ αρχής, αν το ξέραμε ότι ήταν προσπόληση. Το ίδιο έχουμε να απαντήσουμε για τα θέματα ασφάλειας. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια και την πιο έντονη χρήση της τοποθεσίας ήταν αυτές που μας οδήγησαν να αγοράσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου για να υπάρχει ε, πιο κλειστή πρόσβαση, να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά παρόλα αυτά να υπάρχει ευρύ χώρο περιβάλλον και να υπάρχει μια κάποια αίσθηση απομόνωση. Γι' αυτό χρειαζόμασταν και λίγο χώρο περιμετρικά για να μην ε, συμβαίνουν όλα γύρω από το κέντρο συνεδρίων όπως ε, συμβαίνει τώρα που είναι περιτριγισμένο ουσιαστικά το κέντρο συνεδρίων. Για θέματα λοιπόν ασφάλεια, ε, το γεγονό ότι είμαστε στη μέση του πουθενά. Είναι απομονωμένο το μέρο αυτό. Και αυτό ήταν και το σκεπτικό. Αυτό ήταν Ωστόσο ήταν ο στόχος στην επιλογή της τοποθεσίας. Αυτό θεωρώ ότι δίνει χρόνο για περισυλλογή και βγάζει τον κόσμο έξω από το χάος, το καθημερινό. Τα θέματα ασφάλεια νομίζω ότι παραμένουν τα ίδια. Είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε στην τοποθεσία αυτή και ο ενδεχόμενο ε, κακόβουλο που θέλει να επιτεθεί δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πλέον έκτημα σε σχέση με άλλα μέρη. Προφανώς, ναι, στα μέρη αυτά, στην τοποθεσία αυτή γίνονται ε, υψηλού επίπεδου συναντήσεις, όπως για παράδειγμα οι συνεδριάσεις του Προεδρείου που προαπαιτούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Δεν μπορούμε να κάνουμε λοιπόν οποιαδήποτε υποχώρηση σε θέματα ασφάλειας. Η Ένωση Ζων Μονέ. Αυτό το ερώτημα να το απαντήσει η κυρία Ιτσελ, η συναδελφός μου από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας. Εγώ να απαντήσω στον κύριο Αντρέιζεν το εξή. Η νομική διαδικασία για την αγορά και αγοροπολισία ε, οικοπαίδων είναι ότι καταρχάς σας παρέχουμε τις πληροφορίες. Μας προσέγγισε ο ενδεχόμενος πολιτής και όταν μας δοθεί μια πρώτη τέτοια έγκριση ξεκινούμε τις ε, διαδικασίες διαπραγμάτευσης, όπου και καθορίζονται οι όροι της σύμβασης. Στη συνέχεια ερχόμαστε και πάλι σε εσά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης, χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση στην παρούσα φάση και οποιαδήποτε επίπτωση στον προπολογισμό. Και, ναι, όντω το σπίτι που γειτονεύει με το οικόπεδο δεν είναι ικανοποιητικό Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια οικοδομής ε, του κτηρίου και θα ξεκινήσει η ανακαίνιση του κτηρίου αυτού αργότερα μόνο. Είναι πολύ μικρό το σπίτι, 100 τετραγωνικά μέτρα μόνο και θα πρέπει επίσης να ανακαινιστεί ακολουθώντας τις ε, τοπικές οδηγίες για τα κτίρια. Δεν είναι τεράστιο το έργο γιατί δεν θα ταιριάζει άλλωστε και στο περιβάλλον σε ένα μικρό γαλλικό χωριό. Ε, κυρία Ιτσελε, ευχαριστώ πάρα πολύ από τη Γενική Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Οίκου Ιστορίας. Ε, την προηγούμενη χρονιά αναλάβαμε τη διαχείριση του κτηρίου Ζαν Μονέ, που την διαχειριζόταν το κτηρίο, η Ένωση Ζαν Μονέ. Ε, δημιουργήθηκε μια υπηρεσία στη μονάδα του οίκου Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ε, υπήρχε λοιπόν μια διαδικασία που ήταν ε, επίσημη η διακτησία του Ζαν Μονέ. Δημιουργήσαμε μόνιμα προγράμματα, δραστηριότητε για σχολεία, εκπαιδευτικά, για να προωθηθεί η ζωή και η σημασία του Ζαν Μονέ για την ιστοσελίδα τώρα. Υπάρχει ακόμα η ιστοσελίδα της Ένωσης Ζαν Μονέ, αλλά στην παρούσα φάση φτιάχνουμε μια ιστοσελίδα για τη ζωή και το έργο του Ζαν Μονέ στα πλαίσια της υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα διευκρινίσουμε το θέμα ιδιοκτησία. Η Ένωση Ζων Μονέ του χρόνου θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τη δική τη ιστοσελίδα, γιατί στην παρούσα φάση ακόμα υφίσταται η οργάνωση αυτή και ελπίζουμε να συνεχίσουν και αυτοί να διαδίδουν τη σημασία του έργου του Ζων Μονέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βίλαντ. Ευχαριστώ να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις και να προσθέσω κανένα δύο πράγματα, γιατί παρακολούθησα την διαδικασία στο Προεδρείο. Ο Ζαν Μονέ αντιαφισβήτητα είναι προπάτορα και από του ιδρυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να του αφήσουμε να χαθούν, θέλουμε να αξιοποιήσουμε την φήμη του. Γι' αυτό λοιπόν Στην Ένωση Ζαν Μονέ, πολλά από τα άτομα αυτά είναι άτομα ε, από το στενό κύκλο του Ζαν Μονέ, οι οποίοι όμως και αυτοί πλέον είναι κάποιες ηλικίε και δεν μπορούν να συνεχίσουν το έργο αυτό. Χωρίς ε, αυτούς ε, τους εθελοντές δεν θα ήταν δυνατόν να συνεχιστεί το έργο αυτό. Προσπαθεί λοιπόν να διατηρηθούν κάποια εθελοντικά στοιχεία γιατί πραγματικά είναι σε καλή κατάσταση η Ένωση και εκφράστηκε η επιθυμία να συνεχίσουν ε, προγράμματα μετακπαίδευσης για την νεολαία και για άλλους. Και επειδή αυτό το καλλιτέχνημα είναι στη μέση του πουθενά, εντάξει, δεν είναι στη μέση του πουθενά, είναι στην άκρη του πουθενά. 50 χιλιόμετρα από τις Βερσαλίες. Ο Μονέ λοιπόν το επέλεξε το μέρος αυτό σκόπιμα για να μπορεί κανείς να έχει λίγο την ησυχία του. Ακόμα και σήμερα έχει την ησυχία του. Δεν υπάρχει όμως δυνατότητα διανυκτέρευσης. Γι' αυτό λοιπόν θέλαμε να συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε την έκταση αυτή. Το θέμα ήταν κατά πόσον θέλαμε να πάμε 25 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα παραπέρα και να δεν σε ένα πολύ ακριβώς μέρο, ακριβό μέρος. Αυτό λοιπόν ήταν η λογική των τελευταίων 10-15 ε, χρόνων. Γενικά υπάρχει μία τάση ε, λιτότητας και περικοπής εξόδων. Να σας προτείνω να επισκεφτείτε λοιπόν το μέρος αυτό και να το δείτε με την ίδια στα μάτια. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Κανείς άλλος, σχόλια. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται σιγά σιγά το θέμα αυτό, το οποίο και θα καταλήξει σε εμά ε, προφανώς. Ευχαριστώ. Και να περάσουμε στο επόμενο σημείο για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, Αλληλεγγύης για αρρωγή προς την Ελλάδα. Κύριε κυρία Καϊλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αφορά τον περασμένο Φεβρουάριο που στην Ελλάδα, στο νησί της Κρήτης που ξέρετε ότι είναι ο ηλιόλουστο στην Νότια Ελλάδα εκεί έζησαν απρόβλεπτες πολύ σοβαρές καιρικές συνθήκες εξαιρετικά κακό καιρό, εξαιρετικές κακοκαιρίες ε, κυκλώνα που έπληξαν το νησί απρόβλεπτες συνθήκες ε, άγνωστες για την Ελλάδα και φυσικά λόγω της γεωγραφικής θέση ε, της χώρας, αλλά ειδικότερα για ένα νησί όπω η Κρήτη, η τοπική υποδομή δεν ε, είχε προβλεφθεί για τόσο σοβαρέ καιρικέ συνθήκες και η Κρήτη ε, επλήγει από την απώλεια πολλών ανθρωπίνων ζώων. Ε, πέραν των, ζημιών, ε, των υλικών ζημιών, τεράστιες ορεινές περιοχές στους νομούς των Χανίων και τη ρεθύμνη, μπλοκαρίστηκαν, η πρόσβαση στα χωριά ήταν αδύνατη και οι επιτόπου υποδομές και εγκαταστάσει υπέστησαν τεράστιες ζημιές. Ε, πολλές από αυτές τις ζημιές ε, επικεντρώθηκαν στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του νησιού, περιοχές αγροτικές ε, κατά κύριο λόγο που καταστράφηκαν ολοκληρωτικά. Επιπλέον καταστράφηκαν σπίτι των πολιτών. Συνολικά οι άμεσε ζημίες εκτιμάται ότι ανέρχονταν σε 182 εκατομμύρια ευρώ. με το 2% του ΑΕΠ αυτής της περιοχής. Εφαρμοζόντα λοιπόν το συντελεστή 2,5 που προβλέπεται για τέτοιε περιπτώσει, για τι φυσικέ καταστροφέ, η, Επιτροπή υπολόγισε ότι το Ταμείο Ελληνικής θα πρέπει να συμμετάσχει με 4,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων ένα μικρό ποσοστό έχει ήδη ε, καταβληθεί τον Ιούλιο. Ωστόσο, εκκρεμούν 4.500 ε, ε, ευρώ ακόμα για αυτή την ε, περιοχή. Οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να εγκρίνετε αυτό το ποσό, το υπόλοιπο και σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Ευχαριστούμε. Κάποιος σκιώδης που θα ήθελα να σχολιάσει. Κύριε Παπαδημούλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για όσα μας είπε και για τη δουλειά της ε, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή που συνέβη στην Κρήτη. Είναι και αυτή η παιδί της κλιματικής αλλαγής. Η ζημιά είναι πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σημαντική για την οικονομία της Κρήτης. Ε, και η βοήθεια που δίνουμε από το σχετικό ταμείο, όπως προτείνεται στην έκθεση, είναι το 2,5% αυτής της ζημιάς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εγκρίνουμε γρήγορα αυτή την έκθεση και να φροντίσουμε έτσι ώστε να εγκριθεί αυτή η έκθεση και στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου, όπως προτείνεται, έτσι ώστε το γρηγορότερο αυτό το μικρό ποσό να πάει για να ανακουφίσει την περιοχή, καθώς οι δαπάνες για τις επισκευές και τις επιδιορθώσεις έχουν ήδη προχωρήσει με ευθύνη του κράτους μέλους της πατρίδας μου, της Ελλάδας. Ζήτησα το λόγο και για ένα παραπάνω ε, λόγο, για ένα παραπάνω επιχείρημα. Βλέποντας την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε αυτό το ταμείο, διαπιστώνω ότι έχουμε ένα μεγάλο αδιάθετο ποσό, το οποίο μπορεί να φτάσει ενδεχομένως και μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια, που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να επανεξετάσουμε το όριο του 2,5% των ζημιών που αναπληρώνεται από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε γιατί είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις όπου οι πολίτες βλέπουν στη ζωή τους μια έμπρακτη αλληλεγγύη. Αν μπορέσουμε λοιπόν αυτή η αλληλεγγύη να είναι ισχυρότερη, θα είναι καλύτερο για όλους. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για τα κράτη-μέλη, και για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Άλλα σχόλια. Θέλει να σχολιάσει η Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την υποστήριξη της έκθεσης, της πρότασης, συγγνώμη. Ευχαριστούμε. Ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 7η Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι και ότι η έκθεση θα ψηφιστεί στις 25 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ. Πάμε στο σημείο 12, το πρωτόκολλο υλοποίησης της συμφωνίας, της αλληλευτικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου. Κύριε Φερνάνδε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά, κύριε Πρόεδρε. Αυτή η πρόταση συμφωνίας για το νέο πρωτόκολλο δίνει τη δυνατότητα αλίευσης ε, στην περιοχή της Γουινέας Μπισάου. Βασίζεται στις καλύτερες και μεγαλύτερες, ευρύτερες επιστημονικές ε, ε, γνωμοδοτήσεις που είναι δυνατόν να έχει κανείς. Σεβόμαστε την βιωσιμότητα και τη συνοχή με τις λοιπές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά διασφαλίζονται. Όσον αφορά το ζήτημα του προϋπολογισμού υπάρχει ένα οικονομικό αντιστάθμισμα 15 εκατομμυρίων 600.000 ευρώ, εκ των οποίων 11.000 αφορούν την πρόσβαση στους ελευτικούς πόρους για όλες τις κατηγορίες που προβλέπει το πρωτόκολλο. Και μετά υπάρχει ένα ποσό 4 εκατομμυρίων ευρώ για την συνδρομή στην τομεακή ανάπτυξη της αλίας για τη Γουινέα Μπισάου για αυτή την περίοδο που θα ισχύει το πρωτόκολλο. Εγώ θεωρώ ότι το πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει συνεπώς να εγκριθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τη Γουινέα Μπισάου. Ευχαριστώ. Any of the που θα ήθελε να σχολιάσει, κυρία Βαλμίνη. Ε, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι κατά βάση συμφωνώ ε, με τον εισηγητή για αυτή την έκθεση είναι πολύ σημαντική. Θέλω να υπογραμμίσω ότι το νέο πρωτόκολλο υπογράφηκε μετά από ενδελεχή και πολύ ακριβή αξιολόγηση, εκτίμηση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Η αξιολόγηση, η εκτίμηση αυτή αφορούσε και την επίδραση των αποτελεσμάτων του προηγούμενου πρωτοκόλλου. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το ανανεώσουμε πόσο μάλλον που πυρήνα του νέου πρωτοκόλλου είναι η προώθηση τη γαλάζια οικονομία των ζητημάτων βιωσιμότητα. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε 100%. Ευχαριστούμε, κυρία Ιε. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Ο Λιβιέ Σαστέλ παρακολούθησε εκ μέρου του Ζουρινιού τον φάκελο. Απουσιάζει δυστυχώ, οπότε θα σα ενημερώσω εγώ για τη δική του άποψη. Ευχαριστούμε κύριε Φερνάνδες. Ε, με τη θετική μας γνωμοδότηση υποστηρίζουμε τη βιωσιμότητα της αλίας στη Γουινέα Μπισάου και τους ε, σχετικούς τομείς και τις δραστηριότητες. Θα παρακολουθούμε ώστε ο τομεακός αυτός ε, κλάδος να αξιοποιεί πλήρως την βιωσιμότητα των αληφτικών πόρων. Ευχαριστούμε. Πάμε στο επόμενο σημείο. Επόμενο σχέδιο γνωμοδότηση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρωτόκολλο υλοποίηση τη Συμφωνία ε, Εταιρική Σχέση στον τομέα τη Αλία μεταξύ τη Δημοκρατίας, της ε, Λαϊκή Δημοκρατία του ΣΑΤΟΜΕ και Πρίνσιπε και τη Ευρωπαϊκή ε, Κοινότητα. Κύριε Φερνάνδε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία ανανεώθηκε και τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2011 ανανεώθηκε ε, με έναρξη την ημερομηνία αυτή. Ωστόσο, αυτό το πρωτόκολλο δίνει τη δυνατότητα στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλιεύουν στα ύδατα αυτά, στο Σατομί και Πρίνσιπε. Και εδώ έλειψαν υπόψη καλύτερες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σε αφορά τη Διεθνή Οργανισμό για τον Ατλαντικό και αξιολογήθηκαν όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν έκανε τη δική της αξιολόγηση του πρωτοκόλου και των προηγούμενων πρωτοκόλων. Όλα αναλύθηκαν ενδελεχώς. Έγινε διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερομένων. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα που τη δική μα αρμοδιότητα, Επιτροπή Προπολογισμών, το ετήσιο ε, αντιστάθμισμα οικονομικά είναι 840.000 ευρώ, 400.000 ευρώ για την πρόσβαση ε, κατά την περίοδο ισχύω της συμφωνίας και μετά υποστήριξη για την αλληλευτική πολιτική του Σάτομε και Πρίνσιπε ύψους 440.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας. Είναι σημαντικό για τη χώρα αυτή Όλα αυτά με γνώμονα το σεβασμό προς την, πολιτική, την πολιτική του Σάτομε και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ έχω απολύτως θετική γνώμη. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάποιος κοιόδης που θα ήθελε να παρέμβει, να σχολιάσει. Αν όχι, εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίαση. Αλλά να σας υπενθυμίσω πρώτα ότι στις 21 Νοεμβρίου έχει ακυρωθεί η συνεδρίαση και αντικαθίσταται με μια συνεδρίαση στο Στρασβούργο στις 25 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους. I